Ανακοινώσεις. Η κυρία Φραντσέσκα Βαρατσού από τις 28 Φεβρουαρίου έχει αναλάβει καθήκοντα στην Ιταλική κυβέρνηση. κυβέρνηση. Ο κύριος Κλάους Χάινερ Λένε από 1η Μαρτίου 2014 ε, αναλαμβάνει καθήκοντα ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τους συγχαίρω και ενημερώνω σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού ότι σε σχέση με την κυρία Μπαρανσού από τις 28 Φεβρουαρίου για τον κύριο Λένα από την 1η Μαρτίου χειρεύουν οι θέσεις τους. Δυνάμει του άρθρου 74 του κανονισμού μας ε, έχω υπογράψει μία σειρά πράξεων μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και οι πράξεις αυτές θα προσερθούν στα πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης. Και προχωρώ στην ημερήσια διάταξη και τις αλλαγές της ή καλύτερα την